Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων επίση προτείνει την εξή διόρθωση ενός από τα κείμενα τα οποία ενέκρινε το Κοινοβούλιο. Για τον κανονισμό 596 κάθος 2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή κάποιων νομικών πράξεων στην διακανονιστική διαδικασία. Με έλεγχο. Τέταρτο τμήμα και υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος γράφων ε, κομισιών, ε, συμβουλίου κλπ. Δεν πρόκειται να σας τον ε, διαβάσω τώρα. Θα μπορείτε να το δείτε άμεσα στο Sion on Direct και έτσι θα κάνουμε μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου. Περνάμε τώρα στο πρόγραμμα εργασίας, στο οριστική πρόταση του ημερησίας